Κυρίε Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα καλωσορίσω όλου μαζί στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ανάπτυξη. Έχουμε μαζί μας τον Σταφάν Μιστούρα, ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία, τον Στίβεν Μπράιν επίσης, γραμματέα για ζητήματα ανθρωπιστικά και κατεπίγουσα βοήθειας του ΟΗΕ. Also ich äh, Καλωσορίζω λοιπόν μεταξύ μας. Τον ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία, Στάφαν Ντοεμιστούρα, ο οποίος νομίζω τον Φεβρουάριο του 2015 ήλθε τελευταία φορά στην Επιτροπή μας και τον κύριο Στίβεν Μπράιεν, γραμματέα για θέματα ανθρωπιστικών υποθέσεων και συντονιστεί για την κατεπίγουσα βοήθεια. Τα δύο αυτά θέματα προφανώ συνδέονται απόλυτα μαζί τους, μεταξύ τους. Βλέπουμε τι γίνεται στο Χαλέπ τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες ώρες. Καταδεικνύει αυτό πόσο δραματικά είναι τα πράγματα από πολιτικής και ανθρωπιστικής άποψης. Γι' αυτό λοιπόν πείτε μας κύριε Δεμιστούρα, πιστεύετε ότι υπάρχει καν ελπίδα για μια συνευτική διαδικασία ή μήπως η Ρωσία και ο Ασάντ αποφάσισαν να τα ρυθμίσουν όλα στρατιωτικά. Και πάει η ειρηνευτική διαδικασία. Τι συνέπειες θα υπήρχαν και τι θα σήμαινε αυτό και για τον κόσμο και για τη χώρα. Τα προβλήματα δεν διευκολύνονται ασφαλώς, η επίλυση τους δεν διευκολύνεται. Τα ανθρωπιστικά λοιπόν ζητήματα βλέπουμε, τα θέματα των προσφύγων, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ συνεργάζονται στενά στην Συρία, στο Ιράκ, στην Τουρκία, στο Λίβανο, στην Ιορδανία, κοιτώντα πόσο προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χορηγήσει βοήθεια στο Χαλέπι, αν ήταν δυνατόν από πολιτική άποψη να αποστέλουν τα κονβόη βοήθειας. Αυτά φυσικά δεν μπορούμε να τα κάνουμε χωρίς τα Ηνωμένα Έθνη. Και πέρα από το θέμα αυτό, είναι σαφές για μένα ότι μετά τα λάθη που κάναμε εμείς ως κράτη-μέλη το 2015 σε ό,τι αφορά το Ταμείο για τους πρόσφυγες θα πρέπει να αντιληφθούμε καλύτερα ότι μια τέτοια κατάσταση χρήζει, χρήζει πολυμερούς προσέγγισης και συνεργασίας. Δεν μπορούν αυτά να απειληθούν ε, σε εθνικό επίπεδο. Από κοινού μόνο. Μπορεί να ρυθμιστεί και το ε, θέμα της ειρήνευσης και το θέμα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ήμουν εγώ στην ε, αποστολή του Κοινοβουλίου και είχατε δυνατότητα να μιλήσω και με τον μέλλον, μέλλοντα Γενικό Γραμματέα, τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος έχει προσέλθει εδώ στην Επιτροπή μας ως ε, ύπατος εκπρόσωπος για τα δικαιώματα των προσφύγων. Μίλησα πριν από δύο-τρεις ε, εβδομάδες και στη Νέα Υόρκη και να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανακοινώσαμε ανακοίνωσε μάλλον ότι προτίθεται να έρθει και στην Επιτροπή μας. Και ψάχνουμε να βρούμε μια ημερομηνία. Με ενδιαφέρον λοιπόν περιμένω να ακούσω το πώς ορίζετε την, ε, και περιγράφετε την κατάσταση και τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να γίνει. Κύριε Ο'Μπράιεν. Danke, Herr Danke Ich werde auf Englisch reden. Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ, θα μιλήσω στα αγγλικά, αν μου το επιτρέπετε, αλλά μπορώ να απαντήσω στα ε, ιταλικά, στα γαλλικά, στα σουηδικά, στα γερμανικά. Με κάνετε να ζηλεύω, λέει ο πρόεδρος. Όχι καθόλου, δεν θέλω. Ε, λοιπόν, ο κ. Ντεμιστούρα, ήμουν εδώ πριν από ένα χρόνο Και επειδή εσείς έχετε υποστηρίξει εκτενούς τις δράσεις των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα στα όσα συμβαίνουν στο Χαλέπι, με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα, θέλω λοιπόν να σας δώσω πρώτα απ' όλα μια γενική εικόνα των διαφορών σεναρίων τα οποία εμείς μελετάμε. Διότι αυτά μπορεί να μας καθοδηγήσουν στο πώς θα αναλύσουμε τα επόμενα βήματα για την εποχή μετά, αφού τελειώσει το πρόβλημα στο Χαλέπι. Και όπως είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος, για να δούμε τι θα γίνει μετά από την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και εν ώψη και της μεταβατικής φάσης ε, που επέρχεται μια νέα κυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένας νέος γενικός γραμματέας. Να σας δώσω μια εικόνα. Τα Ηνωμένα Έθνη, χάρη σε εσά ε, δεν υπήρξαν αδρανοί Εγώ ξεκίνησα πριν από 26 μήνες και τότε είχαμε γενική ύφεση μετά από το Γενεβή 2. Η εντύπωση που είχαμε λοιπόν εμείς ήταν δραματική και είπαμε πώς θα βοηθήσουμε να προχωρήσει το θέμα της Συρίας και τότε υπόθηκε ότι δεν ε, εκδηλωνόταν κανένα ενδιαφέρον για μια πολιτική λύση παρότι όλοι αναφέρονταν σε πολιτική λύση. Παρεπιπτόντως ε, αυτή την οδό ακολουθήσαμε και μέχρι χθε, ε, για να το πω έτσι, διότι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμή είναι ότι ενώ όλοι ισχυρίζονται και εξακολουθούν να ισχυρίζονται, διότι πολιτικά είναι ορθό να το λέει κανεί, ότι η μόνη λύση είναι πολιτική, σαφώ εντείνονται οι στρατιωτικέ επιχειρήσει οι οποίε αργότερα θα συσκευαστούν σε ένα ωραίο πολιτικό πακέτο ε, Ε, τώρα παρατηρούμε μία αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ε, περιγράφουμε τα πράγματα. Πάμε 26 ε, μήνες πριν από σήμερα, τότε δεν υπήρχε ελπίδα, αλλά εγώ είχα μια διέστηση. Έβλεπα κάτι νέο. Ξέρετε, κάθε κρίση περιέχει και μια ευκαιρία. Και τότε εγώ έβλεπα τον Ντάες Και ε, σκεφτόμουν τότε ότι επειδή τον ΝΤΑΕΣ απειλεί τους πάντες, όλοι θα ενωθούν για να πολεμήσουν τον κοινό εχθρό, τον ΤΑΕΣ και έτσι θα ελύνονταν τα προβλήματα στη Συρία. Λοιπόν, έκανα λάθος κυρίε και κύριοι. Όλοι συνέχισαν να ακολουθούν ε, ε, το δικό του συμφέρον, ενώ ταυτόχρονα επιπροσθέτως μερικές φορές πολεμούσαν τον ΤΑΕΣ. Το επόμενο βήμα λοιπόν ήταν τι θα κάνουμε για να αποφύγουμε τον δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο στη Συρία επειδή κατέληγε να γίνει σαν τη Σομαλία. Ε, θα, θα, έφτανε να ξεχαστεί, να είναι ένα ζήτημα ε, θλιβερό, 200.000 νεκροί, χιλιάδες ε, τραυματίες και πολλοί πρόσφυγες στις γειτονικέ χώρες. Το ζήτημα λοιπόν ήταν πώς θα γινόταν να διατηρήσουμε τη Συρία στην επιφάνεια και εκεί προέκυψε το Χαλέπι. Και κατά παράδοξο τρόπο τα πράγματα πάντα επιστρέφουν στο Χαλέπι, διότι σε τελική ανάλυση το Χαλέπι έχει σημαντική πολιτική, ε, πολιτισμική και συναισθηματική σημασία. Ούτε αυτό λειτουργήσε, διότι τότε το Χαλέπι η μείωση της βίας στο Χαλέπι δεν βοηθούσε τους αντιμαχόμενους τότε. Ε, Ούτε ο Ασάντ βοήθησε τότε, διότι βομβάρτιζε τι γύρω περιοχέ. αλλά η αντιπολίτευση θεώρησε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να δείξει συμβαστικό πνεύμα. Και μετά ήρθε μια νέα πρωτοβουλία, το να μιλήσουμε με του Σύριου, αφού όλοι μα έλεγαν και εμεί λέγαμε η κρίση στη Συρία ε, είναι, πρέπει να επιληθεί μέσω μιας συριακής πολιτικής ε, διαδικασίας. Στη Γενέβη λοιπόν ε, για μεγάλο χρονικό διάστημα συναντηθήκαν πολλές ομάδες όσοι εμπλέκονταν στη Συρία, ειδικότερα τότε η ΜΚΟ, η κοινωνία των πολιτών, τον οποίο τη γνώμη δεν ακούει κανένας όπως ξέρετε στη Συρία. Και γυναίκες φυσικά. Βασική προτεραιότητα για μένα, διότι έχουν την απίστευτη δυνατότητα να ε, είναι πολύ πιο επικοδομητικές από τους άντρες. Ε. Αυτό έγινε με τις διαβουλεύσεις στη Γενέβη, αλλά δεν υπήρξε η κρίσιμη μάζα. Έλειπε το ενδιαφέρον των διαφόρων χωρών ε, να αντιμετωπίσουν τη Συρία ως ένα κοινό πρόβλημα. Και ξαφνικά τρεις παράγοντες έγιναν πραγματικότητα ταυτόχρονα, έτσι όπως γίνεται η ιστορία συνήθως. Μερικές φορές χωρίς να το προκαλέσει κανείς. Ο πρώτος παράγοντας ήταν η προσφυγική κρίση, την οποία γνωρίζετε καλά. Ξαφνικά η Ευρώπη ένιωσε ότι ε, εισέβαλε μια νέα κρίση και απασχόλησε ε, τους, ε, όλους τους πρωθυπουργούς, όλες τις χώρες σε επίπεδο πρωθυπουργών, διότι αποσταθεροποιούσε την Ευρώπη και εξακολουθεί, αποσταθεροποιούσε τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις και επίσης ε, από άποψη ε, υλικοτεχνική αποτελούσε ένα τεράστιο ανθρωπιστικό πρόβλημα. Δεύτερον, κάτι που έλαβε χώρα ταυτόχρονα και ανεξαρτήτως ε, των διαστάμενων απόψεων άλλαξε το παιχνίδι, άλλαξε την εξίσωση η ρωσική στρατιωτική παρέμβαση. Και το τρίτο, ο τρίτος παράγων τον Ντάεσ που ενέτεινε τις δραστηριότητες του όπως ο έμπολα εκμεταλλεύεται την αδυναμία ενός σώματος και επεκτείνεται και ξαφνικά είχαμε επιθέσεις διάφορα ε, γεγονότα και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό αποτέλεσε το καμπανάκι που ξύπνησε την Ευρώπη. Όλες τις χώρες και ειδικότερα τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ρωσία διότι για να εμπλακεί χρειάζεται και μια στρατηγική εξόδου. Και η Αμερική λόγω της πίεσης από εσάς, από τους Ευρωπαίους ουσιαστικά αυτό οδήγησε στο να αποκτήσουν ένα πραγματικό δραστη... Ε, ενδιαφέρον ε, για την Αμερική να εμπλακεί πολιτικά, όχι στρατιωτικά. Ε, και εξού και ο Τζον Κέρι που, και οι προσπάθειές του να προσπαθήσει να απαλύνει την κρίση στη Συρία. Ο συνδυασμός των δύο οδήγησε ουσιαστικά των τριών παραγόντων οδήγησε σε μια σειρά πολύ σημαντικών γεγονότων. Επιτέλους έχουμε μια ομάδα επαφής. Δύο task force, μια ανθρωπιστική και μία για την πάυση των εχθροπραξιών. Είχαμε και κάτι νέο στη Γενέβη, ένα κέντρο επιχειρήσεων, ένα επιχειρησιακό κέντρο όπου συνεργάζονταν οι στρατοί Ρωσίας και ΙΠΑ για να καταλήξουμε σε εκεχηρία, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Είχαμε μια εκεχηρία πραγματικά, μια πάυση του πυρός που διήρξε τρει μήνες. Ποτέ δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό. Το γεγονό ότι τόσες πολλές χώρες και τόσε πολλές εμπόλεμε ομάδες σταμάτησαν, όταν τελικά η Ρωσία και η ΕΠΑ συμφώνησαν την πάυση των εχθροπραξιών, όλοι ηρέμησαν. Αλλά δεν κράτησε πάνω από τρει μήνε. Και μετά η κυβέρνηση της Συρίας θεώρησε ότι ήταν προώρο, ότι δεν είχε νικήσει και η Ανούστρα που είναι τρομοκρατική οργάνωση, εμπόλεμη οργάνωση, δεν ήθελε να έχει υπάρξει εχθροπραξιών. Και αυτό οδήγησε σε άρση της εκεχηρίας. Αλλά για τρεις μήνες ε, σώθηκαν περίπου 11.000 ζωές πιθανότατα. Και όπως θα σας πει και ο Στίβεν Ομπράιον, ένα 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν προσπελάσιμοι στις ε, πολιορκημένες περιοχές, ε, τόσο ε, πολιορκημένες από ε, διάφορες δυνάμεις. Οπότε σταδιακή κατάρρευση. Και αυτό μας φέρνει στη σημερινή κατάσταση. Είχαμε μια προσπάθεια στις 9 Σεπτεμβρίου, την τελευταία στιγμή, στη Γενέβη, από τον Τζον Κέρι και τον Σεργέ Λαυρόφ, και εγώ ήμουν εκεί, μετά τα μεσάνυχτα συζητήθηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση την οποία μπορώ να σας παρουσιάσω αυτή τη στιγμή γιατί ακόμα είναι ζωντανή κατά κάποιο τρόπο αλλά τότε της αμπόταραν δύο γεγονότα. Το πρώτο ήταν η πάυση των εχθροπραξιών και ειδικότερα των βαρτισμών στο Χαλέπι. Δεύτερο, ε, αποχωρισμός της Ανούσρα να, απο, να απομακρυνθεί από τις άλλες ομάδες η Ανούσρα. Η Ανούσρα είναι Αλκάιντα, ναι, έχουν αλλάξει το όνομα, Όπου και τα τσιγάρα αλλάζουν το όνομά τους και, ε, παρότι τα παράγει ιδιαίτερη, αλλά η πραγματικότητα είναι ίδια. Και μετά το τρίτο σημείο που ήταν το πιο ενδιαφέρον για μένα ήταν η... Ε, το σταμάτημα των εχθροπερσών από τη Συριακή αεροπορία. Κανένας βομβαρδισμός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή ως ευκαιρία, πολλά υποσχόμενη, ειδικότερα επειδή εξετάστηκε κάθε λεπτομέρεια. Και αυτό μου έδωσε εμένα πολλέ ελπίδε. Και τότε ήμασταν έτοιμοι να επανεκκινήσουμε τι συνομιλίε για τη Συρία που είχαν ακυρωθεί ήδη τρει φορέ αλλά χωρί κανένα αποτέλεσμα. Διότι η Συριακή κυβέρνηση έλεγε δεν μπορούμε να μιλάμε για μελλοντικό σύνταγμα ούτε για τον πρόεδρο Ασάντ. Και η άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση έλεγε είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε μόνο αν ο πρόεδρο Ασάντ ε, αφήσει τη θέση του, διότι και οι δύο πλευρές πίστευαν πραγματικά ότι μπορούσαν να ελέγχουν τη στρατιωτική πλευρά και δεν ήταν έτοιμη για ειλικρινή διαπραγμάτευση. Δύο γεγονότα οδήγησαν σε κατάρρευση τη 9η Σεπτεμβρίου, που ήταν η μεγαλύτερη στιγμή ελπίδα που είχαμε πρόσφατα. Η επίθεση στην Τεραζόρ από την Αμερικανική αεροπορία, ε, κατά λάθο όπω αναγνώρισαν, μια Συριακή στρατιωτική βάση και μετά αμέσως μια επίθεση που ακόμα διερευνάται όπου ένα φόρτηγα και 20 από τους φίλους μας που ε, συνεργάζονται εκεί, ε, ε, φίλοι μας που συνεργάζονται με τον Ερθρό Σταυρό, έχασαν τις ζωές τους. Εκεί ξεκίνησε η εκστρατεία για το Χαλέπι και εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Να κάνουμε λοιπόν και μια απογραφή της σημερινής κατάστασης. Ξέρετε πως για την ανθρωπιστική κατάσταση δεν μπορώ να αρνηθώ όπως ε, μιλάμε για μια επιτάχυνση των στρατιωτικών ε, των στρατιωτικών ε, επιθέσεων και δεν ξέρω πόσο θα αντέξει ακόμα το Ανατολικό Χαλέπι. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε αυξηνόμενη κίνηση σε στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε κατά τη γνώμη μου είναι τα αποτελέσματα όλων αυτών. Και επίσης δεδομένου ότι έχουμε νέα διοίκηση στην Αμερική και επίσης νέο ε, γενικό γραμματέα του ΟΕΕ Ξέρετε ότι ο Αντώνιο Γκουτιέρες είναι πάρα πολύ δραστήριος και ξέρουμε και πόσο proactive είναι. Αυτό θα επηρεάσει ε, τα όσα θα γίνουν από την αρχή της επόμενης χρονιάς, από 1η και από 20 Ιανουαρίου. Άρα λοιπόν τι περιμένουμε να δούμε. Ενδεχομένως δεν μπορώ να σας πω γιατί μεταξύ της σημερινής ημέρας και της 1 η 20ης η ιανουαριου πολλά μπορούν να συμβούν. Για παράδειγμα, μπορεί να καταρρεύσει το χαλέπι. Μπορεί τελικά να πάρει μια απόφαση η Συριακή κυβέρνηση να πει τελείωσε η μάχη, τελείωσε ο πόλεμος, τώρα θέλουμε να κάνουμε μια ειρηνευτική διάσκεψη. Και παρακαλώ πολύ κύριε Ντιμιστούρα να μας το οργανώσετε. Ωραία, αν φτάσουμε στο σημείο αυτό θα δούμε. Και για να γίνει διάσκεψη ειρηνευτική θα πρέπει να εξασφαλίσει συμμετοχή όλων των μερών και βεβαίως χρειάζεται να εξασφαλίσει και τη δυνατότητα σεβασμού του ψηφίσματος το οποίο ομόφωνα ε, ψηφίστηκε το 2254 που είναι ο δικός χάρτης για μια πολιτική μετάβαση και επίσης μια πολιτική, ε, έναν πολιτικό επιμερισμό της εξουσίας, που να είναι βιώσιμος. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ, ο νεεκλεγής πρόεδρος, δεν γνωρίζουμε τι πολιτική θα ακολουθήσει. Ούτε εσείς ξέρετε, ούτε εμείς και ακόμα δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι ο, ο Υπουργός Εξωτερικών. Έχει όμως κάνει κάποιες δηλώσεις και βασιζόμενοι στις δηλώσεις αυτές έχουμε την εντύπωση πως στόχος του είναι να δώσει πρώτη προτεραιότητα στην μάχη κατά του ISIS. Οπότε δεν νομίζω του Ισλαμικού κράτους. Οπότε δεν νομίζω ότι οποιοδήποτε στις Βρυξέλλες ή στο Παρίσι θα του φέρει αντίρρηση. Ούτε εγώ. Γιατί αν μιλήσει κανείς για οποιοδήποτε άνθρωπο κοινό θα μας πει ότι όχι, δεν θέλουμε ε, που δεν είναι να ξαναβιώσουμε τέτοιες στιγμές όπως αυτές που ζήσαμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελών. Οπότε, εάν πρόκειται κάποια κοινή συμμαχία με τον πρόεδρο Πούτιν έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το Ισλαμικό κράτος στη Ράκα, στη Μοσούλη κατά τη δική μου ταπεινή άποψη βασιζόμενη στο ψήφισμα του ΟΗΕ τότε θα έχουμε κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, είπαμε να δώσουμε τη μάχη για να πολεμήσουμε το Ισλαμικό κράτος. Πώς μπορούμε να, να καταφέρουμε να ιτηθούν Λοιπόν, ένας τρόπος υπάρχει μόνο και αυτό το μήνυμα προσπαθώ να μεταφέρω στη νέα διοίκηση των ΗΠΑ, όπως επίσης και στη Ρωσία, είναι μόνο εάν έχεις ένα καινούριο τρόπο διακυβέρνησης της Συρίας που θα είναι ανοιχτό σε όλους. Γιατί το Ισλαμικό κράτος τρέφεται από τον εκνοβρισμό, την οργή, το θυμό των κοινοτήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται ε, στην διακυβέρνηση της χώρας. Τι έγινε στο Ιράκ. Οι Σουνίτες στο Ιράκ αισθάνθηκαν πως είχαν χάσει τα δικαιώματά τους και γι' αυτό ακολούθησαν τους ρυθμούς του κυρίου Ζαρκάου που ήταν τότε η Αλκάιντα. Αν είχαμε μια διακυβέρνηση του Ιράκ που είχε συμπεριλάβει και τις φυλές και τους Σουνί, τότε ο κύριος Ζαρκάουι θα είχε γίνει μια μικροομάδα που πια έτσι καλώς δεν υφίσταται. Ε, όμως δεν, κάναμε, δεν ε, το επιτρέψαμε αυτό και αντιμετωπίζουμε το Ισλαμικό κράτο σήμερα. Και στην Συρία έχουμε τις περιπτώσεις των μειονοτήτων που αισθάνονται πως δεν έχουν φωνή. Αν θέλει λοιπόν κανείς να ιτηθεί το Ισλαμικό κράτος, χρειαζόμαστε μία πολιτική ε, εξίσωση για τη Συρία που θα είναι ανοιχτή σε όλους ανεξάρτητα με το αν θα βρούμε μια στρατιωτική ή μη στρατιωτική λύση. Σας ευχαριστώ. Κλείνω εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δημιστούρα για τα όσα μας είπατε, για τα όσα μας εξηγήσατε και ελπίζω πως θα πετύχετε. Θα ήθελα τώρα να χαιρετήσω ε, και μια ομάδα νέων ε, πολιτικών από το Ισραήλ και από την Παλαιστίνη που έχει προσκαλέσει το κοινοβούλιο μας. Ο κύριος Ομπράιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε ε, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, όπως επίσης κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Ντιμιστούρα, για μία παρουσίαση ε, γεμάτη πυγμή, ε, απόλυτα τεκμηριωμένη, περιγράφοντας το παρόν και το παρελθόν και ενδεχομένως και το μέλλον της κατάστασης στην Συρία. Και πιο πολύ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την στράτευση με την οποία προσπαθείτε εσείς να βρείτε μια λύση που θα ικανοποιήσει τα αιτήματα του Συριακού λαού. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα που είμαι εδώ και έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω μέσω των επιτροπών σας γιατί είστε ένας ε, βασικός πυλώνας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και μέσω ημών μπορώ να απευθυνθώ στα πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες που εσείς εκπροσωπείτε στα 27 κράτη-μέλη. Γιατί σε τέτοιου είδους παγκόσμια ζητήματα είναι σημαντικό. Ήμουν υπουργό, ήμουν βουλευτής και εγώ δίνω ιδιαίτερη σημασία στο χρόνο ε, που έχω τώρα ως διεθνής ε, δημόσιος υπάλληλος να κάνω τέτοιες ανταλλαγές μαζί σας. Γιατί εσείς μας δίνετε την άδεια να προχωρήσουμε και να δράσουμε κι εσείς και σε εσά πρέπει να λογοδοτήσουμε για τα τεράστια ποσά τα οποία ψηφίσατε εσείς που έχουν πληρώσει τα δικά σας, η δική σας ε, εκλογής για να πληρώσουμε για τις προσπάθειες που κάνουμε. Και πρέπει να σας πω πως η υψηλότερη πολιτική επένδυση είναι αυτή που κάνει κανείς για έκτακτη βοήθεια ανθρωπιστική, για ζητήματα ανθρωπιστικά, για να στηρίξουμε αυτούς που θα θέλαμε να μας στηρίξουν αν είχαν αντιστραφεί οι ρόλοι μας. Και θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω γιατί το κάνετε εσείς για να στηρίξετε το Συριακό λαό. Έχει περάσει πάνω από μία δεκαετία ε, αιματηρής και ε, απίστευτης ε, βίας. Έχουμε δει όλοι τις φοβερές εικόνες με βόμβες οι οποίες βομβαρδίζουν ιατρικά κέντρα, σχολεία, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αγορές, εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους σε όλη τη χώρα και αυτές τις συνεχείς βασανιστικές εικόνες ανθρώπων οι οποίοι έχουν εκτελεστεί, έχουν βασανιστεί, έχουν ακροτηριαστεί, έχουν τραυματιστεί με τον καθημερινό βομβαρδισμό που δεν σταματάει ούτε τη νύχτα. Έχουμε όλες αυτές τις εκθέσεις που ακούμε συνέχεια για χημικά όπλα, για κάθε είδους βόμβα, βόμβα διασποράς, βόμβα ναπάλ, ε, αυτοκτονίες, ε, σνάιπερ, ε, ελεύθερους σκοπευτές, ε, αποκεφαλισμούς, βιασμούς, ε, μεσαιωνικές ολόκληρων πόλεων, ε, τις σε σχολεία, σε νοσοκομεία, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους και πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί. Το προσδόκιμο ζωή, αυτή τη στιγμή στην ε, Συρία έχει πέσει πάνω από 20 χρόνια και τουλάχιστον το μισό του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί. 6,5 εκατομμύρια μέσα στη χώρα, συν μισό εκατομμύριο Παλαιστίνοι πρόσφυγες 5 εκατομμύρια σχεδόν Σύριοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα και το 13,5, τα 13,5 εκατομμύρια που ζουν ακόμα στη χώρα έχουν άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας. 80% των Σύρων ζουν στη φτώχεια και 9 εκατομμύρια περίπου δεν έχουν αρκετά τρόφιμα με τις ελλείψεις σε τρόφιμα και με τις τιμές που αυξάνονται κάθε μέρα. Πουθενά δεν είναι χειρότερη η καθημερινότητα από ό,τι στο Χαλέπι, όπου έχουμε αυτή τη στιγμή μία φοβερή στρατιωτική δύναμη και βία που ασκείται με τρομακτικές συνέπειες. Όπως είπατε κι εσείς, το Χαλέπι έγινε αυτή τη στιγμή ο πυρήνας της κόλασης όπου είναι ανίποτο το πόσο υποφέρει ο κόσμος. Δεν υπάρχουν στο Ανατολικό Χαλέπι ε, νοσοκομεία για να βοηθήσουν όσους ξέφυγαν από το θάνατο. Και ό,τι υπάρχει βομβαρδίζεται μέχρι να εξαφανιστεί. Γίνονται ε, καθημερινά ατέλειωτες μάχες μέσα στην πόλη. Έχουμε ε, επιθέσεις από στρατιωτικά αεροπλάνα, βομβαρδισμούς, ε, ρουκέτες που επιβάλλουν σε όλους να καταλήψουν τη χώρα. Άλλοι παγιδεύονται και δεν μπορούν να μετακινηθούν, άλλοι χάνουν τα σπίτια τους. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να αισθάνεται ο κόσμος ασφαλής. Από τον Ιουλίου 270.000 και αυτό είναι 100.000 παιδιά έχουν παγιδευτεί στο Ανατολικό ε, Χαλέπι λόγω της πολιορκίας που ξεκίνησε η Συριακή κυβέρνηση και η συμμαχίτσα. Εγώ ζήτησα να έρθουν όλες οι πολιορκίες που έχουν γίνει μία από ε, από τα χειρότερα φαινόμενα αυτής της ανηλέητης επίθεσης. Και αντίθετα αυτό που βλέπουμε είναι μία χρήση όλο και μεγαλύτερη της πολιορκίας και όλο και περισσότερους ανθρώπους που πολιορκούνται από την κυβέρνηση της Συρίας. Τέτοια εποχή πέρσι ο αριθμός των πολιορκημένων ήταν 393.700. Έξι μήνες πριν ήταν 486.700 άτομα και σήμερα έχουμε φτάσει 974.080 άτομα. Δηλαδή σχεδόν ένα εκατομμύριο Σύριοι απόψε ζουν υπό πολιορκία. Όπως είπα για τους Σύρους και το είπα στο Συμβούλιο Ασφαλείας δεν υπάρχει τίποτα ε, ε, το οποίο να είναι θετικό για αυτή την πολιορκία, τίποτα που να φροντίζει τους αμάχους, τους βομβαρδίζουν, δεν περνάνε τρόφιμα, δεν υπάρχουν γιατροί, δεν υπάρχουν νοσοκομεία και το μόνο που μπορούν να κάνουν να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν. Είναι μια ε, επιλεγμένη τακτική σκληρή, αδυσόπιτη για να καταστρέψουν ένα πληθυσμό ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και ο χειρότερος, ε, το χειρότερο είναι ότι αυτός ο οποίος θα έπρεπε να προστατεύει τους ίδιους του τους πολίτες ε, δεν το κάνει γιατί όλα αυτά θα έπρεπε τουλάχιστον την ηθική μας συνείδηση να την ταρακουνήσει και να πούμε πως δεν είναι δυνατόν σε μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου να κινδυνεύουμε από την απόλυτη καταστροφή του πληθυσμού. Να έχουμε 100.000 παιδιά παγιδευμένα σε υπόγεια, χωρίς νοσοκομεία που δεν έχουν πού να κρυφθούν. Είναι πρόστιχο είναι αυτή η αδυσόπιτη, ε, το αδυσόπιτο αιματοκύλισμα στο οποίο έχει διολυστήσει η Συρία. Και πραγματικά είναι ανατριχιαστικό να σκέφτεται κανείς ότι αυτό το επίπεδο βίας γίνεται κάτω από τη μύτη μας, μια και υπάρχει μια ελάχιστη ε, δυνατότητα πρόσβασης ε, των διεθνών οργανισμών. Είναι μια σύραξη που συνεχίζεται τόσα χρόνια με τόσες συνέπειες που πραγματικά η παγκόσμια συλλογική συνείδηση θα έπρεπε να να ε, κλαίει για το γεγονός ότι επιτρέψαμε να συμβεί κάτι τέτοιο. Τα μέλη λοιπόν ε, του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να σκεφτούν το εξή. Αυτό η σύραξη στο εσωτερικό της Συρίας έδειξε τα χειρότερα στοιχεία του ανθρώπινου γένους, αλλά σε ορισμένε περιπτώσεις έδειξε και το καλύτερο. Εγώ πήγα στη Συρία, έχω πάει στην διευρύτερη περιοχή και μίλησα σε πάρα πολλού Σύριου, οι οποίοι εξακολουθούν να ελπίζουν ακόμα και είδα τη γενοδορία οικογενειών στο Ιράκ, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στο Λίβανο ε, και παντού αλλού που μοιράζονται το λίγο που έχουν με αυτούς τους ανθρώπους και είδα τι κάνουν οι παόμικρον στη Συρία, οι Συριακές και είδα τι κάνει η Αραβική Μισέλινος, την ανέφερε και ο Στέφαν, είδα τι κάνουν οι, οι, εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, σε κλινικές, σε σχολεία που πεθαίνουν και αυτοί πολύ συχνά γιατί έχουν συστρατευτεί έτσι ώστε να σώσουν τους συμπολίτες τους. βλέπω τι γίνεται και με το δικό μου προσωπικό, το προσωπικό του ΟΗΕ, τι ανθρωπιστικέ οργανώσει που κάθε μέρα, κάθε ώρα διακινδυνεύουν για να πάνε βοήθεια σε αυτού που χρειάζονται περισσότερο. Ξέρετε πω ο ΟΗΕ και οι ενώσει αυτέ εργάζονται αδιάποκα κάθε μέρα για να σώσουν τους Σύριους είτε μέσα στη Συρία είτε προσφέροντας βοήθεια στο εξωτερικό. Παρόλο που οι προϋποθέσεις είναι απίστευτες και φέτος καταφέραμε να βοηθήσουμε 5,8 εκατομμύρια ανθρώπους με τρόφιμα κάθε μήνα. Και αυτή η βοήθεια πηγαίνει μέσω προγραμματισμού και ε, μέσω, περνώντας τα μέτωπα από τη Δαμασκό και μέσω της Ιορδανίας και μέσω της Τουρκίας. Και επειδή έχουμε αυτές τις διασυνοριακές επιχειρήσεις εδώ και δύο χρόνια, ο ΟΗΕ κατάφερε να, κάνει πάνω από, να στείλει πάνω από 420 κομβόι ε, συνοριακά, δηλαδή πάνω από 4 την εβδομάδα, με φάρμακα για 9 εκατομμύρια ανθρώπους, με εμβόλια για 2 εκατομμύρια ανθρώπους, με τρόφιμα για 3 εκατομμύρια ανθρώπους, πολλά σε μηνιαίο, σε μηνιαία βάση και βοήθεια που δεν είναι... Ε, ε, τρόφιμα, αλλά είναι ε, ήδη υγιεινής και νερό σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχουμε στείλει βοήθεια σε πολλά κομμάτια, στο Χαλέπι, στη Λατάκια, στη Χαμά, σε πολλές περιοχές από την ε, Τουρκία και σε άλλες πόλεις της Συρίας από την Ιορδανία. Πρέπει εσείς να ξέρετε πως η δική σας βούληση και οι δικέ σας, ε, τα δικοί σας πόροι κατάφεραν να μεταφραστούν σε μια πραγματική ανθρωπιστική βοήθεια που έσωσε εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό γιατί η κλίμακα είναι τέτοια, αυξάνεται συνέχεια και οι δικές μας προσπάθειες βέβαια βοηθά και τις ΜΚΟ, τη Διεθνής και άλλους οργανισμούς που προσπαθούν να βοηθήσουν εκατομμύρια Σύριου στο εξωτερικό. Προσπαθούμε και δια αέρος. Έχουμε μια αεροδιακομιδή που ε, αυτή τη στιγμή έκανε 153 ε, ε, αποστολές έτσι ώστε να καταφέρει να στείλει 61.000 ε, δελτία ε, καλάθια με τρόφιμα, ε, δηλαδή 5,7 κυβικά μέτρα από τρόφιμα, από είδη υγιεινής, από νερό και σε αυτό θα πρέπει να συμπληρώσω πως καταφέραμε και 61.500 μερίδες φαγητό με τον ίδιο τρόπο και πρέπει να σας πω πως ε, χτες ο ΙΕ η Ερυθράη Μισέλνος, η Αραβική Μισέλνος και ο Ερυθρός Σταυρός κατάφεραν να στείλουν στη Μηδία, στο Ζαμπεντάνι ε, και στην Κουφρία τρόφιμα για άτομα μετά από χιλιάδες ώρες διαπραγματεύσεων και με έναν συντονισμό έτσι ώστε να καλύψουμε τουλάχιστον τις ανάγκες 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Και πρέπει να σας πω πως ήταν ηρωικές οι ομάδες μας επί τόπου που γύρισαν το βράδυ στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα έχοντας παραδώσει αυτά που πήγανε που ήταν από τα σπάνια καλά νέα που είχαμε από αυτή την πλημμυρίδα αρνητικών ενστάσεων, νέων, γιατί κάθε μήνα στέλνουμε τέτοιου είδους αιτήματα στη Συριακή κυβέρνηση και κάθε μήνα μας στέλνουν γραφειοκρατικά εμπόδια γιατί εμείς δεν μπορούμε να παραδώσουμε. Εγκρίσεις που έρχονται καθυστερημένες, εγκρίσεις που έρχονται με περιορισμό στους δικαιούχους, εγκρίσεις με το να έρθουν τα φορτηγά στις αποθήκες, εγκρίσεις που δεν έρχονται για τη διαδρομή, ιατρικά, υλικά που δεν μπορούμε να παραδώσουμε και μετά όλα αυτά που συμφωνούμε δεν μας επιτρέπουν να τα κάνουμε επιτόπου. Και ξέρετε πως ήταν ελάχιστα αυτά τα κομβόι που κατάφεραν να φτάσουν ε, φέτος το καλοκαίρι. Ξέρετε πως οι Σύριοι οι οποίοι εγκαταλείπουν τη βία και τον πόλεμο θα ρισκάρουν οτιδήποτε πάνω σε φουσκωτά και σε σαπιοκάραβα για να πάνε οπουδήποτε. Και ξέρετε το 2016 πολλοί από αυτούς που πνίγονται στη Μεσόγειο είναι Σύριοι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να αιτηθούν άσυλο χωρίς καμία διάκριση. Και για να λύσουμε α, τα προβλήματα αυτών των προσφύγων υπάρχει βάρος για την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε πως ο συναλλικός αριθμός αυτών στην Ευρώπη οχριά σε σχέση με αυτούς που έχει υποδεχθεί η Τουρκία, το Ιράκ, ο Λίβανο και η Ιορδανία. Ένα τέταρτο του πληθυσμού της Λιβύης αυτή τη στιγμή είναι πρόσφυγες από τη Συρία. Και για τη Γαλλία, να σας πω, το Ηνωμένο Βασίλειο πως είναι αν είχαμε το αντίστοιχο 1 τέταρτο θα είχαμε 15 με 17 εκατομμύρια πρόσφυγες. Και αν ήταν το ίδιο ποσοστό στην Ουγγαρία ή στη Σλοβακία θα ήταν 2 με 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Εάν κάνουμε αυτή την απλή Έχουν φάει ε, τα λεφτά τους, οι οικονομίες τους, τα κορίτσια παντρεύονται νωρί για να μπορούν να φύγουν ενώ θα έπρεπε να πηγαίνουν σχολείο και έχουν τραυματιστεί ψυχολογικά και σωματικά. Ξέρετε πως ε, τα παιδιά στο Χαλέπι θα πήγαιναν σχολείο το Σεπτέμβριο. Δεν πήγαν. Και αντίθετα αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μέσα στα συντρίμια παιδιά τα οποία παίρνουμε με μαντωμένα ρούχα και τα στέλνουμε σε νοσοκομεία που βομβαρδίζονται, που δεν μπορούν ούτε να κοιμηθούν, ούτε να παίξουν, ούτε να διαβάσουν. Ένα από τα τέσσερα σχολεία στη χώρα δεν λειτουργεί. Πάνω από 52.000 δάσκαλοι εγκατέλειψαν τη δουλειά του. Πάνω από 2 εκατομμύρια παιδιά εγκατέλειψαν το σχολείο. Και να σα πω πω άλλα 2 εκατομμύρια πρόκειται να εγκαταλείψουν γιατί συνεχίζεται ο αδυσόπιτος αυτό απέσιο πόλεμο, 100.000, χιλιάδες χιλιάδες παιδιά είναι απάτριδες και τα έχει εγκαταλείψει η οικουμένη και δεν έχουν μέλλον. Και τι μέλλον θα έχουν, είναι ορφανά, πεινάνε, είναι αμόρφωτα. Ποιο είναι το μέλλον αυτής της χώρας, τι θα κάνει η επόμενη γενιά, είναι χαμένη. Χρειάζεται να τους βοηθήσουμε και χρειάζεται να βοηθήσουμε και τις κοινότητε που τους υποδέχονται. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια ολιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει ε, όλη την γάμα των ανθρωπιστικών τους αναγκών, δηλαδή από τους εκτοπισμένους που είναι στις γειτονικέ χώρες, από τους πρόσφυγες που μετακινούνται και θα πρέπει την επανεγκατέσταση τους σε άλλες χώρες να τη στηρίξουμε. Αυτό το Κοινοβούλιο στις 6 Οκτωβρίου και στις 24 Νοεμβρίου ενέκρινε ψηφίσματα και τα ψηφίσματα αυτά είναι σημαντικά αλλά θα πρέπει να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Γιατί επιτρέψτε μου να είμαι ειλικρινής. Θέλουμε καλύτερη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής απόκρισης για τη Συρία και την περιοχή. Θέλουμε να ε, ξαναβρούμε ε, το, τη δύναμή μας από την αρχή της χρονιάς που τη χάσαμε. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος της βίας, πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος και χρειάζομαι χρειάζεται όλα τα μέρη να εξασφαλίσουν πως θα έχουμε μία ανθρωπιστική πρόσβαση η οποία δεν θα αντιμετωπίζει κανένα πρόσκομα και μία άμεση διακοπή αυτών των μεσαιωνικών πολιορκιών που βασανίζουν ανηλέητα όλα αυτά τα εκατομμύρια αμάχους. Γιατί αν δεν λύσουμε τις πολιορκίες δεν θα κάνουμε τίποτα. Και καλό όσους έχουν επιρροή σε οποιοδήποτε μέρος ε, σε αυτή τη σύραξη. Καλό εσά το Κοινοβούλιο να κάνετε ό,τι μπορείτε αυτή την παράλογη, αυτό το παράλογο κύκλο βία να το διακόψουμε, να σταματήσει πια το αιματοκύλισμα στην Συρία. Η Ευρώπη θα πρέπει να δείξει ηθική ηγεσία και να αναλάβει υποχρέωση όχι μόνο στα λόγια για να προστατεύσει του πιο ευάλωτου, αυτού που έχουν ανάγκη, αυτού που αντιμετωπίζουν βιοπραγίε, εγκλήματα και απερίγραπτη ε, απερίγραπτο πόνο. Θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη τις διαφορές μας και η διεθνής κοινότητα με μια φωνή να ζητήσει να σταματήσει αυτή η ντροπή που μας βαραίνει όλους για πάντα και επιτέλους να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνευση στη Συρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπράιν. Και νομίζω ότι μας δώσατε μια στιγμή περισλογής για την πολιτική αποτυχία και την ανθρωπιστική καταστροφή και τα πολλαπλά θύματα. Από πλευρά του Κοινοβουλίου παρακολουθούσαμε την κατάσταση διαρκώ, αλλά μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε κάνει και κάτι παραπάνω. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να αφιερώσουμε κάποια σκέψη για την πολιτική αποτυχία. Και τώρα σήμερα ασφαλώ σκεφτόμαστε το χαλάκι και το όσο συμβαίνουν εκεί. Αναφέρατε, κύριε Ομπράιαν, τα όσα συμβαίνουν στη, με τους πρόσφυγες και στην στενή μας γειτονιά. Ήμουν, υπήρξε αποστολή στο Λίβανο, στον που πήγαν ε, συνάδελφοι. Είδαμε πώς έχει κατάσταση λοιπόν στις γειτονικέ ε, χώρες και δραστηριοποιήθηκαμε για τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική βοήθεια σε ό,τι αφορά την ε, εκπαίδευση των νέων παιδιών των νέων. Γιατί ξέρουμε ότι είναι σε κατάσταση επικίνδυνη, κινδυνεύουν να χάσουν όλη την παιδική του ηλικία και το μέλλον του χωρί εκπαίδευση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι πάρα πολύ σοβαρέ αυτέ παρατηρήσει. Το θέμα λοιπόν που ανακύπτει τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το παρελθόν. Διάφοροι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο και να ξεκινήσουμε. Έχουμε ω τώρα. Έχουμε μόνο 35 λεπτά στη διάθεσή μας. Να ζητήσω λοιπόν τους συναδέλφους να μην μιλήσουν παραπάνω από λίγα λεπτά ο καθένας. Ο κύριος Πρέντα είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους ε, δύο προκεκλημένους, τον κύριο Τεμιστορα και τον κύριο Μπράιν, για τις παρεμβάσεις τους. Έχω δύο παρατηρήσεις να κάνω. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τα όσα είπε ο κύριος Δεμίστουρα για μια πολιτική λύση. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό θα πρέπει να συμβεί. Έχουμε ένα θέμα διαφορά απόψεων σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία τη Ρωσία. Γιατί η Ρωσία δεν βρίσκεται στη Συρία βάσει ψηφίσματο του ΟΗΕ. Α, κλήθηκε προ βοήθεια από τον Ασάντ. Ε, έχει κάνει επιθέσει και σε άλλε περιοχέ. Αυτή η έλλειψη λοιπόν αξιοπιστίας είναι ακόμα πιο οξυμένη γιατί πρόκειται για έναν, μια χώρα η οποία μπλοκάρει τη λήψη αποφάσεων στον ΟΗΕ και έτσι λοιπόν αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και πόσο μάλλον ε, μετά την ανάληψη των καθήκοντων του κυρίου ε, Τραμπ. Ε, αυτή η κατάσταση λοιπόν η πολιτική θα συνεχιστεί όσο η Ρωσία συμπεριφέρεται με τον ίδιο ελεύθερο τρόπο σε ό,τι αφορά το διεθνέ δίκαιο. Και αυτό είναι που βαραίνει. Είναι μια ευθύνη που θα πρέπει να λάβει η Ρωσία και θα πρέπει να την καλέσει προ την κατεύθυνση αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την παρέμβαση του κ. Ομπράιαν, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μα παρουσίασε και είμαστε πολύ περήφανοι στην Ευρώπη που, που θέλησαμε να διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θέλουμε λοιπόν ως Ευρώπη βασικά να διαδραματίσουμε ανθρωπιστικό ρόλο, αλλά αυτό δεν ε, λειτουργεί ασφαλώς πάντα. Βλέπουμε στις ειδήσει τις εικόνες από το Χαλέπι και βλέπουμε ότι η κατάσταση η ανθρωπιστική δεν χαρακτηρίζεται από παρέμβαση της ε, διεθνού κοινότητα και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Οι Ρώσοι, οι στρατιώτε είναι αυτοί που τελικά βοηθούν τους αμάχους και δυστυχώς με λείπει το αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η πρόεδρος, η κυρία Μακέφεν, ο κύριος Νόιζερ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας. Εγώ συμμετείχα στην αντιπροσωπεία στο Λίβανο και μιλήσαμε με άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται σε ομάδες του ΟΗΕ και θα πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικό το έργο του ΟΗΕ στο Λίβανο. Ερωτώ λοιπόν, σε τι βαθμό το πρόγραμμα, το περιφερειακό πρόγραμμα για τους πρόσφυγες σε χρηματοδοτείται και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούν τι δεσμεύσει του, γιατί υπήρχε θέμα χρηματοδότηση τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τρόφιμα. Αναγκαστικά μειώθηκαν τα τρόφιμα προς τους πρόσφυγες. Δεύτερο ζήτημα. Χρειαζόμαστε καλύτερη υποστήριξη της κυβέρνησης του Λίβανο, γιατί μετά από δυόμιση χρόνια επιτέλους έχουμε εκ νέου μια κυβέρνηση και είναι τόσο μεγάλη επιβάρυνση του Λιβάνου που θα πρέπει να φροντίσουμε τη σταθεροποίηση αυτό. Το τρίτο σημείο αφορά την τρέχουσα κατέσταση στο Χαλέπι. Δυστυχώς όλα οδεύουν προς στρατιωτική λύση. Σε τι βαθμό λοιπόν ο ΙΕ προτίθεται να βοηθήσει σε περίπτωση τακτικής επέμβασης ε, με ανθρωπιστικό τρόπο ε, τον, ε, τους, α, αμάχους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στίβεν, θα με θυμάσαι, είχαμε διπνήσει μια φορά μαζί όταν ε, έκανα την έκθεσή μου ως ειδικό απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασίλειου για το Σαχέλη, είναι σαφές ότι είναι βιβλικών διαστάσεων η καταστροφή η οποία εκτίλησε τόσο μιλάμε από τις ε, ρωσικές και ε, συριακές δυνάμεις. Πριν από πέντε χρόνια στο Κοινοβούλιο είχα ζητήσει μία no-fly zone, μία ζώνη με απαγόρευση πτήσεων, που δεν έγινε τότε. Είμαι περήφανο που το ζήτησα τότε, αλλά δεν υπήρχε πολιτική βούληση τότε πολύ απλά. Τρει ερωτήσει έχω να κάνω. Καταρχά, έχετε σκεφτεί καθόλου στα πλαίσια του ΟΗΕ να επικαλεστείτε το 377 του ΟΗΕ για την ένωση ε, του Συμβουλίου του ΟΗΕ για την καταδίκη της Ρωσίας σε ό,τι αφορά την επιβολή ενός ρονευτικού σχεδίου ή μήπως αυτό αποτελεί ευσεβή πόθο. Σε ό,τι αφορά τον μέλλοντα πρόεδρο Τραμπ, πέρα από την προτεραιότητα για την απολέμηση του ISIS, αναρωτιέμαι μήπως θα κάνει κάποια συμφωνία με τον Πουτίν για την Συρία έναντι Ουκρανίας, σε ό,τι αφορά τον ανθρωπιστικό διάδρομο από το Χαλέπι. Ένα από τα βασικά θέματα που μας ανησυχούν στην Ευρώπη είναι ότι μεταξύ των ε, πραγματικών προσφύγων θα κρύβονται και πολλοί τζιχατιστές από την, ε, το Ισλαμικό κράτος και ούτω καθεξής. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη δεν θα είναι τέτοια προέλευση και θα είναι πραγματικά άμαχοι. Ιδιαίτερο τώρα που η Ράκα και η Μοσούλη πιέζονται παράλληλα και συνεχίζονται και η καταδίωξη των δυνάμεων του Ντάες. Τελευταία ερώτηση. Ε, φαίνεται ότι υπάρχει ένας πόλεμος διαντιπροσώπου μεταξύ Σεϊτών και Σουνιτών. Είναι πραγματικά εφικτή η μελλοντική διατήρηση της Συρίας ως ένα κράτος. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν ε, ισχύει. Μην ξεχνάμε ότι ήταν ε, Γάλλοι υπεύθυνοι για τη χάραξη των συνόρων μεταξύ Συρίας, Ιράκ κτλ. Μήπως έχει έρθει η ώρα να τα ανακαλέσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Καστάλντο από το EFTD και μετά θα ξεκινήσουμε με τους ομιλητές από πλευρά των ομάδων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, πρεσβή κύριο Ντιμιστούρα και τον ε, αναπληκτή γραμματέα Μπράιν για την εκτενή παρουσίαση. Ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις, ε, ειδικότερα προς τον κύριο Ντεμιστούρα. Πρώτα απ' όλα, ένα σχόλιο για τον ρόλο της Τουρκίας. Ε, αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαδραματίζει ένα ρόλο όχι τόσο επικοδημητικό αλλά καταστρεπτικό όπως φαίνεται. Ακούσαμε πολύ σοβαρές διακήρυξεις από τον Ερντογάν, ο οποίος αμφισβητεί και τα σύνορα της συνθήκης των Σευρών ε, εκφράζει ότι θέλει να παίξει ένα ρόλο και να επηρεάσει τα πράγματα τόσο όσον αφορά τη Μοσούλη στο Ιράκ και όσον αφορά την απελευθέρωση της Ράκα κάνει προσπάθειες να αποτελέσει κομμάτι των, ε, ε, της καταστροφής της ισορροπίας σε διάφορα σημεία. Είναι μια στάση σοβαρής αντιπαράθεσης και με τους Κούρδους και ειδικότερα τους Σύριους Κούρδους. Ήθελα λοιπόν να μου το σχολιάσετε όλο αυτό και δηλαδή πώς βλέπετε τι αποτελέσματα θεωρείτε ότι θα έχει αυτή η παρέμβαση της Τουρκίας στη Συρία και ειδικότερα για τη Ράκα. Δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με την νίκη του Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Πώς πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε ακούσει δηλώσεις που δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι επιθυμεί να συνεννοηθεί με τον Πούτιν και ενδεχομένω να υπάρξει κοινή στρατιωτική παρέμβαση του χρόνου όταν ο Τραμπ αναλάβει πλήρω τα καθήκοντά του μετά από τη μεταβατική περίοδο. Αυτό θα έχει επιπτώσεις ήδη από τώρα ενώ αναμένουμε να καταλάβουμε κατά πόσο οι κινήσεις της Αμερικανικής Διοίκησης ε, θα γίνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ναι, συγγνώμη, δεν είχα δει την κυρία Λοτήλ ε, ως συντονίστρια των Πρασίνων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για τι παρουσιάσει Την περασμένη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετήσαμε ένα ψήφισμα για τη Συρία ένα μεγάλο του οποίου αφορούσε το πώς θα προετοιμαστούμε για την κατάσταση μετά από τις εχθροπραξίες. Και σας ευχαριστώ κύριε Μιστούρα για τα όσα είπατε, ότι θα πρέπει να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών στη Συρία, η διασπορά, οι πρόσφυγες, αλλά και οι γυναίκες. Όλοι θα πρέπει να συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Ε, που θα οδηγήσουν, ελπίζουμε, σε μια κυβέρνηση χωρί αποκλεισμού στη Συρία. Σε αυτή τη διαδικασία πολιτική μετάβαση, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει τα πράγματα κάπω αλλιώ ή κάπω διαφορετικά ή να κάνει περισσότερα πράγματα. Επίση ο κύριος ε, Ομπραϊάν ε, περιέγραψε όλα τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράττονται στη Συρία και το Συμβούλιο Ασφαλείας αναφέρεται σε πιθανή παραπομπή στο Διεθνές ποινικό δικαστήριο. Ποια είναι η δική σα ε, άποψη για τη δημιουργία ενό δικαστηρίου ειδικού για τη Συρία. Δεν είναι βέβαια η καταλληλότερη στιγμή καθώ οδεύουμε προ μια κεχηρία, αλλά ήθελα να ακούσω ποιε είναι οι σκέψει σα από αυτού του ζητήματο. Ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε του ομιλητέ των ομάδων. Ε, θυμηθείτε το χρόνο, γιατί θέλουμε να λάβουμε και απαντήσει. Οπότε παρακαλώ μην επαναλαμβάνετε πράγματα που έχουμε ήδη ακούσει. Ξεκινάμε με το ΕΛΚΑ. Ο κύριο Αντάκτασον. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ομπράιον και κύριε Ντεμιστούρα για τις παρουσιάσεις σας, πολύ ενδιαφέρουσες και πλήρες. Καθημερινά έχουμε έναν σουηδόφωνο ε, στην Επιτροπή μας, ε, οπότε θα μιλήσω στα σουηδικά για να ε, κάνω την ερώτησή μου. Είπατε λοιπόν ότι, ότι το ίσις μπορεί να το νικήσουμε μόνο αν υπάρξει μια καινούρια κυβέρνηση η οποία θα συμπεριλαμβάνει και θα λαμβάνει υπόψη όλες τις διάφορες ομάδες της χώρας. Πείτε μας δύο λόγια παραπάνω. Γιατί όταν συναντιόμασταν με εκπροσώπους μειονοτήτων στην Συρία και παραδέθηκα και στη Δαμασκό συναντήθηκα με τις χριστιανικές ομάδες και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε έντονη ανησυχία. Τι θα γίνει αν κάποια μέρα εξαφανιστεί ο πρόεδρος Ασάντ. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε να φροντίσουμε να συνεχίζουν να προστατεύονται αυτοί που προστατεύονται υπό το σημερινό καθεστώ. Δεύτερο ζήτημα, δεύτερη ερώτηση, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη παταγώδη αποτυχία τη πολιτική σε όλα τα επίπεδα και κυρίω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ πιστεύετε λοιπόν ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει ξανά έναν ενεργό ρόλο στην κατάσταση αυτή, η οποία στην προσεφάση δεν κατέχεται από τη Ρωσία και από άλλους φορείς. Ευχαριστώ η κυρία Βαλενσιάνο, η πρόεδρος της Υποεπιτροπής Ανθρωπινών Δικαιωμάτων, η Ελένη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για όλες τις προσπάθειες που έχετε κάνει και θα ήθελα και να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες τις οποίες έχετε καταβάλει. Η σημασία αυτή της προσπάθειας πολλές φορές δεν φαίνεται στο ε, αποτέλεσμα που πετυχαίνουμε, αλλά παρόλα αυτά αναγνωρίζεται από εμά. Έχω και για τον κύριο Μπράιν μια ερώτηση και για τον κύριο Τιμιστούρα. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για πολιτική λύση γιατί έχουμε τουλάχιστον ένα χρόνο που μιλάμε γι' αυτό, όταν στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα καθαρά καταστροφικό σενάριο, ε, σενάριο στρατιωτικό, ε, καταστροφής ε, αμάχων. Το είπατε στο τέλος, αλλά θα ήθελα να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Και για τον κύριο Μπράιαν ήθελα να ρωτήσω το εξή και θα είμαι πολύ ευθύς. Πώς το αντέχετε. Πώς αντέχετε να είστε στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών προσπαθώντας να, να σώσετε ζωές ανθρώπων που γνωρίζετε και παράλληλα να αντιμετωπίζετε την απόλυτη έλλειψη προτάσεων λύσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Πώς γίνεται να κάνουμε τα δύο αυτά παράλληλα. Ευχαριστούμε πολύ, Ευχαριστώ. Είχα κάποιε ερωτήσει προς τον Στίβεν. Θα θυμάστε ότι εγώ ήμουν υποψήφιος για Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ε, το 2006 ε, απέναντι στον Πάνκι Μουν και ο λόγος που ήθελα να το κάνω ήταν για να μεταρρυθμίσω τα Ηνωμένα Έθνη, το οποίο η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Από το κακό στο χειρότερο πάει και ζητώ συγγνώμη που το λέω. Είναι εντελώς ένας αναποτελεσματικός οργανισμό ο οποίο απλά κάθεται, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Είτε θα μεταρρυθμίσουμε λοιπόν τα Ηνωμένα Εθνή, είτε θα τα κλείσουμε. Δεν μπορεί ο φορολογούμενο τη Ευρώπη να βάζει τόσα λεφτά στα Ηνωμένα Εθνή τσάμπα. Εμεί συχνά χρησιμοποιούμε τα Ηνωμένα Εθνή ω ε, έναν ε, οργανισμό αρρωγή. Ε, όλα είναι αδρανή αυτή τη στιγμή. Όταν αναλάβει καθήκοντα ο πρόεδρος Τραμπ ε, είπε ότι θα ξανακοιτάξει το όλο ζήτημα και εγώ κάθομαι εδώ και μου φαίνεται ότι συζητάμε για το Άμλετ αν θα γίνει ε, πρίγκιπας της Δανίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατό, το ΝΑΤΟ δεν ξέρουμε πού θα οδεύσει, τα Ηνωμένα Έθνη είναι αναποτελεσματικά και ο Τραμπ λέει ότι δεν θα έρθει σε αντιπαράθεση με τους Ρώσους Ε, στο θέμα της Συρίας ε, και ότι θα συνεννοηθεί με τους Ρώσους και θα καταλήξει κάποια, θα συνέψει κάποια συμφωνία. Πολλά κινούνται λοιπόν αυτή τη στιγμή και αυτή η κινητικότητα μας δίνει την ευκαιρία να αποφασίσουμε με ποια πλευρά θα, ε, θα συνεργαστούμε ώστε να βρούμε μια αποτελεσματική λύση ειρηνευτική για την περιοχή. Αλλιώς απλά καθόμαστε και αποφασίζουμε ε, διάφορα πράγματα ενώ ε, ε, βλέπουμε διαδοχικές καταστροφές. Ξέρετε, τα Ηνωμένα Εθνή υποφέρουν όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορούνται για διάφορα πράγματα ενώ ουσιαστικά εθνικές πρωτεύουσες με τις αποφάσεις που λαμβάνουν. Ξέρετε, υπό τον Κόφι Ανάν τα Ηνωμένα Έθνη ήταν αποτελεσματικά, όχι όπως με τον Πανκιμούν, ναι. Αλλά αυτό που λέτε προσβάλλει του εργαζομένου ε, στα Ηνωμένα Έθνη και στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών κρίσεων, ξέρετε, όλοι αυτοί ε, κινδυνεύουν τις ζωές τους ε, για να κάνουν ό,τι μπορούν. Ε, κυρία Σάκα, τον, από του φιλελευθέρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τους δύο προσκεκλημένους μας που ήλθαν και μας ε, μίλησαν για την τεράστια δυσκολία στη δουλειά σας και νομίζω ότι μας σε αυτά που είπε ο κ. Δημιστούρα για την πλήρη απουσία της Ευρώπης. Αυτό ελπίζω να το επιλύσουμε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ομπράιν για την σαφήνεια και την ξεκάθαρο πνεύμα με τον οποίο μίλησε. Και νομίζω ότι επικρατεί μια ντροπή και ένα θυμό τεράστιο, ανίποτο, για την βία που χρησιμοποιείται και για την ε, διασταυρωμένη σχέση μεταξύ του καθεστώτος του Ασάντ και του Ισλαμικού κράτους. Όσοι προειδοποιούν ότι χωρίς τον Ασάντ ε, δεν θα είχαμε τζιχάντ, ε, να δουν πού βρισκόμαστε. Το να χρησιμοποιούνται η δικαιολογία ε, αυτή λοιπόν για να βομβαρδίζονται νοσοκομεία και σχολεία είναι ό,τι χειρότερο έχουμε τα τελευταία χρόνια. Και είναι πάρα πολύ κοινικό ότι λένε κάποιοι ότι υπάρχουν όταν μιλάμε για βία, ε, στη βία. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε όλο και πιο πολύ και πιο μεγάλη ηγεσία στον κόσμο, αλλά σε διαφορά τη Συρία χρειαζόμαστε και ανθρωπιά και πολιτική, πολιτική κυρίω ηγεσία. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν και του δύο σας, ποια τρία βασικά ζητήματα θα ήταν τα σημεία τα οποία θα προβάλλετε ω προτεραιότητε από την Ευρώπη σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και Παντσέρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ντεμιστούρα και τον κύριο Μπράιαν για την παρουσία τους εδώ και για τα όσα ε, κάνουν ε, υπό συνθήκες πολύ δύσκολες και ε, δεδομένων των συνθήκων κάνουν ό,τι μπορούν φυσικά. Κατά την απόψή μου συμβαίνει το εξή. Έχω την εντύπωση ότι η ηθική συνείδηση είναι κάτι που θα μείνει αμετακίνητο αν η πολιτική είναι ανεπαρκής, αν υπάρχουν στρατηγικές διαφορές στην περιοχή ή όπως ε, στην ευρωπαϊκή περίπτωση ουσιαστικά υπάρξει αδράνεια, απουσία. Πιστεύω ότι η εξέλιξη των ανθρωπιστικών ε, ζητημάτων ε, σχετίζεται στενά με το γεωπολιτικό πλαίσιο, το οποίο πλαίσιο δυστυχώς έχει αλλάξει ριζικά και ταχαίως τον τελευταίο καιρό. Για να δούμε τα πράγματα όπως έχουν, σήμερα. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για το Ανατολικό Χαλέπι. Η ρωσική παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική. Αυτό αποτελεί πλέον γεγονός. Και το τρίτο στοιχείο, το οποίο δεν συζητήσαμε, βλέπω ότι η υποστήριξη προς τους ε, επαναστάτες έχει αποδυναμωθεί. Η Τουρκία έχει μειώσει τη βοήθειά της, οι Ηνωμένες Πολιτείες επίσης, το ίδιο και η Σαουδική Αραβία για διαφορετικούς λόγους ο καθένας η Τουρκία διότι έχει μια νέα σχέση με τη Ρωσία όπως υπόθηκε οι Ηνωμένε Πολιτείε για τον Τραμπ, η Σαουδική Αραβία, γιατί έχει άλλα μέτωπα ανοιχτά. Και η ερώτηση που θέλω να θέσω είναι η εξή. Δεδομένου του πλαισίου αυτού, για να αποφύγουμε απλά εμεί να καθόμαστε και να κοιτάμε ε, και για να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να να σκεφτούμε κάποιες λύσεις προβλέποντας ε, τι μορφή θα έχουν και μία από αυτές τις λύσεις αναμφίβολα θα ήταν το πώς εμείς θα διαμορφώσουμε την τελική μορφή της Συρίας. Ε, κατά πόσο θα διατηρηθεί η εδαφική ακαιρεότητα ή αν όπως πιστεύω εγώ είναι προτιμότερο να μην διατηρηθεί. Το λέω διότι έχω την εντύπωση ότι θα υπερισχύσει η νεοαμερικανική ιδέα της προτεραιότητας και ο στρατηγός ε, Πενχέας είπε ότι δεν υπάρχουν προτεραιότητες ε, όσον αφορά την επέμβαση στη Συρία. Εμείς θα πρέπει να κινηθούμε προς αυτή την οδό το πιθανότερο, αλλά αν αυτή η ιδέα του καθορισμού προτεραιοτήτων δεν συνοδευτεί από μια προσαρμογή στο νέο πλαίσιο που θα έχουμε στην ε, Σύρια, πιστεύω ότι όλα τα ανθρωπιστικά εγκλήματα τα οποία αναφέρουμε δεν θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε θα πρέπει λοιπόν να συνδυάσουμε το ανθρωπιστικό ζήτημα με το νέο πολιτικό πλαίσιο το οποίο προσπαθούμε να καθορίσουμε. Thank you. Mr. Ευχαριστώ κύριε Σκορονμίγκε. Ε, to... Πρώτη ερώτηση προς τον κύριο Τζεμιστούρα. Φήμες άκουσα από την Ουάσιγκτον ότι οι μυστικές υπηρεσίες ε, Αμερικής και Ρωσίας ε, συνεργάζοντας στη Ρωσία, για, στην Συρία για να ε, προκαλέσουν στρέβλωση. Γιατί αυτό δεν είναι προς το συμφέρον, όσο γίνεται δεν είναι στο συμφέρον των μυστικών υπηρεσιών. Και ήθελα να σχολιάσετε. Και κατά δεύτερον, οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες σχόλια εκτός μικροφώνου. Επαναλάβατε, επαναλάβατε παρακαλώ. Επαναλαμβάνω. Άκουσα φήμες από την Ουάσιγκτον ότι αμερικανικές και ρωσικές μυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται για να ε, διαστρεβλώσουν για να σταματήσουν αυτή τη συνεργασία και την συνόηση μεταξύ Ρωσίας και ε, Αμερικα... Αμερικής. Αν δεν υπήρχε ανθρωπιστική βοήθεια, θα είχε σταματήσει και καιρό ο πόλεμος. Η ανθρωπιστική βοήθεια είναι αυτή που προ... αναβάλλει την έλεξη του πολέμου. Μετά τον πόλεμο θα πρέπει να δοθεί η ανθρωπιστική βοήθεια, όχι παράλληλα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κόμες. Καλώς ήλθατε στην Επιτροπή μας, κυρία Ντεμιστούρα Στάφαν. Είπατε ότι μια λύση για την Συρία θα περιλάμβανε μια λύση και για τους Σουνίτες. Αυτή η πολιτική για του σουνίτε μπορεί να γίνει με τον Ασάντ, πιστεύετε. Δεύτερη ερώτηση. Ο μελλοντικό πρόεδρο, ο Τραμπ και με τι σχέσεις που έχει σκοτεινέ με τη Ρωσία και με την Τουρκία. Και πώς μπορούν να επιληθούν όλες αυτές οι αντιφάσεις και είμαι από αυτούς που είναι εξοργισμένοι και ντρέπονται ιδιαιτέρως για τις φρικαλαιότητες της ανθρωπιστικής κατάστασης. Πιστεύω ότι δεν αρκούν αυτά που κάνουμε από ανθρωπιστικής άποψης. Ή γιατί τίθεται θέμα δεοντολογίας, ηθικής και πολιτική ηγεσία. Τι χρειάζεται λοιπόν από την Ευρώπη, ερωτώ. Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη για να κάνετε για όχι μόνο να τραυματιστεί ο πόλεμος, αλλά και για να επικρατήσει η ειρήνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τέλος ο κ. Φρόιντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα σχολιάσω το οτιδήποτε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο προσκεκλημένους για την ε, τεράστια αυτή δουλειά που κάνετε. Μισή ερώτηση έχω να κάνω ουσιαστικά, γιατί πιο πολλοί έθεσαν ήδη τα ερωτήματα που ήθελα να θέσω. Τελευταίο ομιλητή και πάντα έτσι γίνεται. Αλλά η Άννα έθεσε το θέμα και ήθελα να τονίσω και αυτό που είπε ο κ. ότι τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη. Όποια και αν είναι ωστόσο η λύση, πολιτική, στρατιωτική. Ο πρόεδρο Ασάντ θα παραμείνει στην εξουσία. Αυτό θεωρώ ότι είναι πέρα κάθε αμφιβολίας. Αυτό όμως πάντα αμφισβητούτα μέχρι πριν από ένα-ενάμιση χρόνο μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με τον Ασάντ. Ε, πολλοί λένε ότι όχι, να φύγει πρώτα ο Ασάντ και μετά βλέπουμε. Η πραγματικότητα όμω πλέον είναι ότι θα παραμείνει στην εξουσία. Αυτό τι θα σημαίνει για τι διαπραγματεύσει μα για την ε, κυβέρνηση ενότητα συμπερίληψη, όπω τον αναφέρετε, το Inclusion Government. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ να κάνω μια ερώτηση, λέει η κυρία Μακέβαν. Από ό,τι φαίνεται θα πέσει το χάλα επί τι επόμενε ώρες Βλέπουμε και τα ανακοινώθεντα τύπου τα σχετικά. 60.000 άτομα, 16.000 άνθρωποι φεύγουν από το Χαλέπι. Ακούσαμε σήμερα το πρέπει που πάνε, περνάνε από δρόμους του ΟΗΕ, ανθρωπιστικής βοήθειας, ε, κινούνται μέσω του Ασάτ. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους για να είναι ασφαλείς αυτοί οι άνθρωποι, τα γυναικόπαιδα. Τι γίνεται ή πλέον όλα είναι στα χέρια της Ρωσίας και της Συρίας. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει πρώτα στο λόγο. Ο κύριος Ομπράιαν, ο κύριος Ομπράιαν λοιπόν και μετά να ακούσουμε και το πολιτικό σκέλος ε, για την αλλαγή του καθεστώτος στο μεγάλο αυτό ερώτημα που τέθηκε. Ο κύριος Ομπράιαν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αισθάνομαι πραγματικά ότι και εσείς ανησυχείτε και επιδεικνύετε αλληλεγγύη με το λαό της Συρίας όσο περνά ε, την, την παρατεταμένη ε, περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης. 80% των 90 εκατομμυρίων ε, που χρειάζονται υποστήριξη για να τα βγάλουν πέρα, για να επιβιώσουν, προκύπτουν από ανθρωπογενείς καταστροφές και συγκρούσεις. Στη Συρία βλέπουμε λοιπόν την πιο βίαιη και πιο έντονη τέτοια σύγκρουση. Η Εμένη και το Νότιο Σουδάν ασφαλώς δεν υστερούν και πολύ δυστυχώς, να απαντήσω στα ανθρωπιστικά πιο πολύ για τα πιο περίπλοκα τα αφήσω το λόγο στον συνάδελφο, στον Στέφαν Δεμισούρα. Με ρωτήσατε συγκεκριμένα, ο κύριος Νόιζερ προφανώς έχει δίκιο ότι θα πρέπει να δράξουμε αυτή την ευκαιρία για να αντιπλασιάσουμε την υποστήριξή μας προς το Λίβανο με τη νέα κυβέρνηση που έχει πλέον ε, αναλάβει τα καθήκοντά της για να έχουμε μεγαλύτερη σύνδεση με τα μέσα τα οποία μπορούν να πετύχουν υποστηρίξη προς τον λαό του Λιβάνου. Γιατί πραγματικά αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Ένα τρίτο του πληθυσμού της χώρας είναι άτομα τα οποία προκύπτουν και έρχονται από εσωτερική μετατόπιση και μετακίνηση. Βλέποντα λοιπόν τον Λίβανο και τον πρόγραμμα το οποίο είναι καλά καταρτισμένο από την υποστήριξη του Λιβάνου, από το τουλάχιστον που α, ανέλαβε ο ΙΕ και η εταιρή του. Έχουμε μία μόνιμη επιτροπή των ε, Ηνωμένων Εθνών μεταξύ υπηρεσιών. Περιλαμβάνει αυτό ταμεία και προγράμματα του ΟΗΕ, αλλά και όλων των άλλων φορέων, παγκόσμιες ΜΚΟ, Παγκοσμία Τράπεζα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι κοιτάμε όλη τη Συρία, τις γειτονικέ χώρες. Πώς γίνεται η χρηματοδότηση έγινε και συνέδρια για τη Συρία και αυτό ασφαλώς θα καθορίσει για τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να τα αναγνωρίσουμε όλα αυτά και να τα, κατασχε... καταρτήσουμε ως σχέδια για τα επόμενα χρόνια να βγει και ένας προπολογισμό για τις άμεσες ανάγκες, τις κατεπίγουσες ανάγκες του επόμενα έτη. Αυτά έχουμε το πρόγραμμα 3RP όπου περιλαμβάνεται μια διαρκής ανθρωπιστική βοήθεια για το πού μπορούμε να παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Όχι μόνο για να επιζήσει ο κόσμος, αλλά για να μπορέσει να ευεμερίσει. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας και τις γνώσεις μας. Αυτά θα τα συζητήσουμε. Τα συζήτησαμε μάλλον το Μάιο του φετινού έτου. Ήταν το πρώτο σχετικό συνέδριο που οργανώθηκε στην ιστορία του ΟΗΕ για την χρηματοδότηση του πρόγραμμα e Είναι 53%. Όπως ε, ήθιστε στον ΟΗΕ στην καλύτερη περίπτωση είναι μισή χρηματοδότηση από πλευρά του ΟΗΕ. Στην καλύτερη περίπτωση το τονίζω αυτό. Και να πω το εξή πριν από 18 μήνε. Εδώ και 18 μήνες εστιαζόμαστε στο θέμα αυτό. Στο εξή, ότι δεν έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε δημόσιο χρήμα από κανέναν, ακόμα και αν διαδραματίζουμε πολύ σημαντικό ανθρωπιστικό ρόλο. Πρέπει να τα κερδίσουμε τα χρήματα αυτά, να πείσουμε τις κυβερνήσεις και όλους εσάς ότι τα χρήματα αυτά, τα οποία είναι χρήματα του φορολογούμενου, ότι τα αξίζουμε. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να, είμαστε, να είναι το έργο μας τέτοιο επίπεδο, ώστε να θεωρείται ότι αξίζει να επενδύσει κανείς σε αυτό. Και ότι είναι πραγματικά κορυφαίας ποιότητας και ότι αξίζει να επενδύσουμε σε αυτό. Αυτό τι σημαίνει όταν λέμε 55%, 45% των πόρων προέρχεται μάλλον 45% των πόρων χρειάζεται για να υποστηρίξει την επιβίωση και την ευημερία των ανθρώπων αυτών, όταν τους σώσουμε με το καλό. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανθρωπιστική διάσωση, 43% είναι η χρηματοδότηση, πιο χαμηλή. 2,49 δισεκατομμύρια του προγράμματος από τα 4,51 δις. Ελπίζω έτσι να καταλαβαίνετε γιατί ύψος ε, πόρων μιλάμε. Αλλά η κυρία Σχάκε, η οποία δυστυχώ μόλις έφυγε, ε, ζήτησε να της πούμε τις τρεις προτεραιότητες μας. Χρήματα, προφανώς. Αλλά να σας εξηγήσω πώς διαμορφώνεται αυτό. Να απαντήσω όμως αυτά στην ερώτηση του κ. Τάνοκ και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπω κ. Τάνοκ για το no-fly zone, για την ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Τέθηκε και ένα ερώτημα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο χθε σχετικά. Ω ανθρωπιστική δύναμη του ΟΗΕ, ασφαλώς ποτέ δεν θέλουμε να καταρριφθεί μία πρόταση σε ό,τι αφορά τις ανάγκες του κόσμου, σε ό,τι αφορά όμως τη ζώνη απαγόρευση πτήσεων. Να θυμόμαστε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό Κανείς δεν αμφιβάλλει για το πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Αυτό για δύο λόγους. Καταρχάς, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ ακριβό. Είναι πραγματικά η τελευταία ίστατη λύση. Υπάρχει δηλαδή α, Υπάρχει ε, ε, ε αεροπορική ε, από αέρος ε, αποστολή τέτοιων πακέτων και βλέπουμε ότι οι μαχητές της, του Ισλαμικού κράτους έχουν όπλα τα οποία φτάνουν σε κάποιο ύψος. Πρέπει να πετάνε λοιπόν πάνω από το ύψος αυτό και παρόλα αυτά να παραμένουν ανέπαφα τα αγαθά. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος προσέλκυσης του κόσμου σε μια ζώνη απαγορευτής πτήσεων, γιατί φυσικά αποτελεί πόλο έλξης αυτό. Και εκτός και αν μπορούμε με όλα τα μέσα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των ανθρώπων αυτών, τελικά κινδυνεύουμε να μεταφερθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη ζώνη και να μην μπορούμε να τους ε, να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά τους. Άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί δεν απορρίπτουμε την πρόταση αυτή ολοκληρωτικά, αλλά χρειάζονται έξι εβδομάδε ε, ε, πτήσεων και εναλλαγή πτήσεων για να φτιάξουμε ένα κόμπο. Γι' αυτό λοιπόν. Ε, αυτή είναι η αντιστοιχία. Για να μπορέσουν να μεταφέρονται τα αγαθά που χρειάζονται. Για τα εγκλήματα πολέμου τώρα και το ερώτημα που τέθηκε. Και εγώ το λέω και ο Γενικό Γραμματέα και ο κ. Ντεμισούρα το λέει. Υπάρχει και πολιτική βούληση των 193 κρατών όπου πιστεύουμε. Και να σας διαβεβαιώσω ότι συλλέγονται αθλητικά στοιχεία. Αλλά αυτό συνήθω ξέρετε συμβαίνει μετά την ολοκληρώση μια σύγκρουση. Είναι λίγο δύσκολο να γίνουν όλα αυτά κατά τη διάρκεια όσο ακόμα εκτελήσεται η σύγκρουση. Και αυτό θα ισχύσει μεταξύ άλλων και για του 20 οδηγού φορτηγών που χάσαμε πριν από κάποιε εβδομάδε σε ό,τι αφορά τον ανθρωπιστικό διάδρομο από το Χαλέπι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αν δεν το κανονίσει αυτό ο ΟΗΕ, φυσικά ε, θα υπάρχει ο κίνδυνο ότι δεν θα συνάδει με το διεθνέ δίκαιο, που ουσιαστικά θα καλέσουμε τον κόσμο να φύγει, αλλά δεν μπορούμε πάλι να εξασφαλίσουμε την ασφαλεία του. Δεν ξέρουμε πού θα πάει δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα φτάσουν με ασφάλεια εκεί που είναι να φτάσουν την ε, ασφάλεια και τη ζωή του κόσμου. Γιατί ο κόσμο έχει δικαίωμα να πάει όπου θέλει. Δεν ε, μπορούμε να του καθοδηγήσουμε υποχρεωτικά σε κατάβλισμου. Και ένα άλλο θέμα για το Ιράκ, όπου προσπαθούμε να κάνουμε ένα εξάρτητο ε, έλεγχο από πλευρά του ΟΗΕ. Είναι πιο αμερόληπτο ο ΟΗΕ σε σχέση με μια οποιαδήποτε άλλη οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Έτσι το τώρα για τα άλλα ερωτήματα. Πρώην συνάδελφο, ε, ο οποίο έθεσε μία ερώτηση για το τι, γιατί ασχολούμαστε με τον ΟΗΕ. Πρέπει να πω πω Εγώ δεν αφιέρωσα την πολιτική μου, ολόκληρη την πολιτική μου καριέρα σε κάτι το οποίο θεωρώ άχρηστο και πραγματικά θαυμάζω αυτό που είδα στον ΟΗΕ που είναι η δυνατότητα να βρίσκουμε θέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν το μάγιστο ε, ελάχιστο παρανομαστή και όχι τον κατώτατο. Καταλαβαίνετε οποιαδήποτε δημόσια οποιοδήποτε δημόσιο οργανισμό τέτοιου είδου είναι μια μεγάλη γραφειοκρατία με όλο και περισσότερου κανόνε. Και ε, όπω και εσεί, για παράδειγμα, έχετε προσθέσει κανονισμού όταν παρουσιάστηκαν προβλήματα χωρί να αφαιρέσετε άλλου, το οποίο σημαίνει περισσότερη γραφειοκρατία, η οποία πολλέ φορέ μου δημιουργεί εκνευρισμό. Γιατί και εγώ προέρχομαι εκτό από τον πολιτικό χώρο και από τον ιδιωτικό κλάδο και πολλέ φορέ αντιμετώπισα προβλήματα με τη γραφειοκρατία. Όσο για την προσωπική μου προσέγγιση, εμείς ξεκινήσαμε στο δικό μου οργανισμό και στη δική μου διεύθυνση να κάνουμε περικοπές, κάνουμε μια αξιολόγηση και είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται συνήθως σε δημόσιους οργανισμούς όπου κανείς δεν περιμένει να βρει πως χάνει το μισθό του, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και αυτό. Και ο προπολογισμό μου για το 2017 σε κάποιες περιπτώσεις προχώρησε σε πολλές μειώσεις. Και δυστυχώ αυτό συμβαίνει <laughs> όταν η αγορά την οποία εξυπηρετούμε ε, αυξάνεται συνέχεια. Καταλαβαίνετε πως οι υποθέσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που χειρίζομαι από 120 εκατομμύρια ανθρώπων έφτασε στα 135 εκατομμύρια και τα 80 εκατομμύρια πρώτη προτεραιότητα έγιναν 92 εκατομμύρια και φτάσαμε να έχουμε ανάγκη 50 δισεκατομμύρια από 22 δις. Γιατί, γιατί στους 18 αυτούς μήνες αυξάνθηκαν οι κρίσεις, οι πόλεμοι και στο παρελθόν είχαμε να κάνουμε με επεισόδια φυσικών καταστροφών και τώρα έχουμε με μακροπρόθεσμες σειράξεις που είναι ανθρωπογενείς. Δεν έχω άλλο χρόνο. Λοιπόν, να πω στα γρήγορα πως θα ζητήσω να αναγνωρίζετε πως εμείς προσπαθούμε να είμαστε ε, επενδυτικής, ε, επενδυτικά ε, αξιόλογοι, το οποίο σημαίνει πως εσείς θα πρέπει να δείξετε στράτευση, να δείξετε οργή και να έχουμε και κάποιες θετικές επιταγές ε, έτσι ώστε να έχουμε αρκετή επιρροή και από τη δική σας πλευρά για να βελτιώσουμε τα πράγματα επί τόπου και να στηρίξουμε και την αναπτυξιακή βοήθεια όσο και την ανθρωπιστική. Και μπορώ να διαβεβαιώσω τον συνάδελφο που το είπε πως η ανθρωπιστική βοήθεια λέει δημιουργεί όλα τα προβλήματα στη Συρία. Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά για να σώσεις μια ζωή. Τελεία και παύλα. Και τέλος, επειδή αυτή τη στιγμή πέφτει το χαλέπι, έχουμε 16 με 22.000 ανθρώπους σε μετακίνηση. Κάποιοι μπαίνουν στο δυτικό χαλέπι, όχι απαραίτητα σε περιοχές που προστατεύονται από τον ΟΗΕ, αλλά και σε άλλες περιοχές, τις οποίες αυτή τη στιγμή έχει η Συριακή κυβέρνηση. Προσπαθούμε και εκεί να είμαστε παρόντες, έτσι ώστε να φροντίζονται και οι άνθρωποι αυτοί σωστά, αλλά είναι χαοτική η κατάσταση, δεν μπορώ να σας το εξασφαλίσω. Φοβάμαι πως ο πόλεμος δημιουργεί χάος και εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι διερμηνείς μας έδωσαν και επιπλέον χρόνο. Οπότε και ο κύριος Δημιστούρα να απαντήσει σε ερωτήσεις αυτές. I will... Ευχαριστώ. Έχετε το πολύ 10 λεπτά. Ωραία, λοιπόν, θα είμαι τηλεγραφικός ή θα προσπαθήσω τουλάχιστον. Πρώτα απ' όλα, η αξιοπιστία της Ρωσίας ε, είναι ένα ζήτημα που τίθεται όσον αφορά τη λύση. Δεν θα μιλούσα για αξιοπιστία ή όχι, θα έλεγα συμφέροντα μάλλον. Και ε, ε, λέγοντας αυτό, βασίζομαι στην υπόθεση ότι όταν έλαβε χώρα η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας, ε, ουσιαστικά αυτό σήμαινε εμπλοκή στη Συρία, την οποία δεν θέλουν να διαιωνίσουν. Δεύτερον, και εδώ βασίζομαι στις δικές μου συνομιλίες μαζί τους, ε, αναζητούν αυτή τη στιγμή μια στρατηγική εξόδου. Με τα λόγια του Colin Μπάουελ, θυμάστε τι, άφησαν πίσω τους οι ΙΠΑ στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και πώς χρειάστηκε να βρουν μια οδό διαφυγής. Είναι καλή πρόταση τώρα αυτή για τη Συρία για τα επόμενη 20 ετία με τον ανταρτοπόλεμο που θα συνεχιστεί πιθανώς σε αγροτικές περιοχές με τα προβλήματα με τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέι, το Κατάρ, τα Εμμυράτα με τόσο κόσμο εντός της Ρωσίας ε, που θα είναι, είναι Σουνίτες, ε, Μουσουλμάνοι και ταυτόχρονα αναμένεται να συμμετάσχουν ε, στην ανοικοδόμηση της Συρίας με τι χρήματα. Όλα αυτά μας οδηγούν στο εξή. Όταν μου λένε ότι δεν τους συμφέρει καθόλου να παραμείνουν εκεί, τους πιστεύω. Τους ενδιαφέρει να βρεθεί μία λύση πολιτική μια πολιτική λύση που να βασίζεται είναι δυνατόν και γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε. Θα πρέπει να είναι, δυνατόν λοιπόν σταθερή και η μόνη σταθερή λύση είναι μια κυβέρνηση οικουμενική που να περιλαμβάνει όλες τις πλευρές και να βασίζεται ε, στο ψήφισμα 2244. Πλησιάζει η ώρα, διότι ε, όταν μιλάμε για ε, ε επιτάχυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα έρθει κάποια στιγμή όπου ο πόλεμος θα έχει κερδιθεί, αλλά αυτή θα είναι μια πύριος νίκη. Χρειάζεται να συνεχιστεί η πορεία της χώρας, να ανοικοδομηθεί η χώρα, να προστατευτούν τα σύνορα, να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει σταθερότητα και ότι δεν θα ξαναεμφανιστεί ένα τάσσα από το πουθενά. Εγώ θεωρώ ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας είναι αξιόπιστες. Ε, απόψη στρατηγικού σχεδιασμού. Δεν είμαι λοιπόν αγαθός, απλά πιστεύω ότι αυτό που μου λένε σε τελική ανάλυση είναι πολύ αληθές. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να κληρονομήσουν μια κατακρεματισμένη, διαλυμένη Συρία. Θα το, πρέπει να το τεστάρουμε δηλαδή, αλλά ε, φυσικά αλλά έρχεται η ώρα. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα για τη χρηματοδότηση για τους πρόσφυγες, το απαντήσατε. Την υποστήριξη προς το Λίβανο, εγώ ήμουν πέντε χρόνια στο Λίβανο, μόνο μπορώ να το υποστηρίξω μπορώ. Ο Λίβανος έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες για να απορροφήσει ε, το αντίστοιχο των 100 ε, εκατομμύριων προσφύγων στην Ευρώπη. σε μια χώρα όπου η βοήθεια από του προσφέρουμε αποτελεί καθήκον για μα. Κατά πόσο είναι δυνατή ακόμα μια πολιτική λύση είναι φυσικά. Ξέρετε, όταν το λέω μπορείτε να μου πείτε ότι ονειρεύομαι. Ε, όλοι σκεφτόμαστε ότι η λίστα είναι στρατιωτική. Ωστόσο, η απάντηση είναι ότι ναι, εντείνονται οι στρατιωτικέ επιχειρήσει, αλλά καμία στρατιωτική λύση δεν μπορεί να νομιμοποιηθεί, να είναι αξιόπιστη, πιστευτή και να παραμείνει σταθερή χωρί πολιτική λύση. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μας θα πρέπει να συμμετάσχουμε ενεργά ε, στο άμεσο μέλλον για την υλοποίηση του 2254 ε, μετά από την κατάρρευση του, στο, της πόλης ε, στο Χαλέπι διότι θα συνεχιστεί ενταρτοπόλεμος για τα επόμενα 5-6 χρόνια. Κάτι που δεν αξίζει στη Συρία, δεν θα υπάρξει καμία ανοικοδόμηση και θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα στη χώρα. Η ουσία λοιπόν είναι πια ότι έρχεται η ώρα όπου θα χρειαστεί να διαπραγματευτούμε και που θα γίνει και η διαπραγμάτευση μεταξύ Ρωσία και Ασάτ και δεν έχει γίνει ακόμα. Τότε θα δούμε πώ έχουν τα πράγματα. Όταν έρχονται στη Γενέβη λένε δεν πρέπει να αγγίξουμε τίποτα ε, εκτό από να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνική ενότητα. Τι σημαίνει αυτό να ε, βάλω εσά ω Υπουργό Γεωργία και εσά ω Υπουργό ε, για ε, κάποιο άλλο τομέα ή απλά να έχουμε μια κυβέρνηση οικουμενική που να περιλαμβάνει τους πάντες. Εκεί θα δούμε πώς έχουν πραγματικά τα πράγματα. Ε, ξέρετε, η Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, ε, ε, ε το Συμβούλιο Ασφαλείας συγγνώμη, των Ηνωμένων Εθνών είναι πραγματικό Συμβούλιο Ασφαλείας και με τα δύο του ψηφίσματα τελευταία δεν δεν έχει αποκλείσει τη δυνατότητα του να υπάρξει ειρήνη. Ασκηπίες είναι αυτά τα ψηφίσματα και όλα αυτά συμβάλλουν ώστε το πρόβλημα της Συρίας να μην πέσει σε δεύτερη μοίρα και να θεωρείται δεδομένο. Οι μελλοντικέ πολιτικές του Πρόεδρου Τραμπ δεν μπορώ να αναλύσω αυτή τη στιγμή. Οι προτεραιότητες του τις έχει εξηγήσει ο ίδιος προφορικά προσωρινά φυσικά, κατά κάποιο τρόπο, απλά έχει κάνει κάποια σχόλια. Οπότε πιστεύω ότι θα τα συζητήσει αυτά με τη δική του ομάδα, αφού θα την έχει συζητήσει. Και ελπίζουμε ότι κάποιο θα το βοηθήσει να καταλάβει ότι πράγματι μπορεί κανεί, ε, θα πρέπει να. ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Ρωσία για να καταπολεμηθεί τον ΤΑΣ. Αλλά μετά από την ήττα του ΤΑΣ θα πρέπει να υπάρξει μια πολιτικά οικουμενική λύση. Αλλιώς η κατάσταση θα επιδεινωθεί. Η Συρία θα γίνει μια βιώσιμη, ενοποιημένη χώρα ή θα κατακαιρματιστεί. Εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω εργαστεί ως ειδικό ε, απεσταλμένος τόσο στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, την εποχή που το Ιράκ και το Αφγανιστάν ε, ζούσαν αυτά που ζει σήμερα η Συρία. Δηλαδή ήταν η τραγωδία της εποχής. Και θυμάμαι εκείνη την εποχή και στις δύο χώρες τέθηκε το ζήτημα του μήπως ο κατακρεματισμός θα ήταν μια καλύτερη λύση. Στο Ιράκ, για παράδειγμα, στο Βορρά έχετε τους Κούρδους, δύο ουσιαστικά κουρδικές οντότητες στο Βόρειο Ιράκ. Έχετε το κέντρο, βόρειο κεντρικό κομμάτι, οι Σουνίτες και οι Αμπάρκοι και μετά η Σιητική περιοχή. που μοιάζει να μην βρίσκεται στην ίδια χώρα. Αν δει κανεί τι διαφορέ, ο τρόπο που ντύνονται οι δραστηριότητέ του και ούτω καθεξή. Ε, τελικά όμω κάτσαν όλοι και είπαν καλύτερα να μείνουμε ω μία χώρα γιατί αλλιώ ανοίγουμε το κουτί τη Πανδώρα. Το ίδιο συνέβη και στο Αφγανιστάν μεταξύ Μπαρτζάνη Σαρίφ και Τζάλα Λαμπάρ, ε, δηλαδή του Νότου και του Βορρά. Μερικοί είχαν προτείνει τον διαχωρισμό και τελικά οι ίδιοι Αυγανοί είπαν όχι. Θέλω να πιστεύω και ε, το υποστηρίζω ως ιδέα ότι η Συρία και αυτό ακούω από κάθε σερό και την αντιπολίτευση και τους ε, φιλοκυβερνητικούς ότι η Συρία πρέπει να παραμείνει μια ενιαία χώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική αποκέντρωση αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε και να αναγνωρίσουν και αυτοί στο τέλος αυτή της φρικτής ε, διαμάχης ότι τα δεδομένα στη χώρα έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιείται η τοπική ε, ε, αυτοδιοίκηση. πιστεύω ότι όμως το μαχισμός της χώρας δεν θα πρέπει να λάβει χώρα. Η Τουρκία έχει 900 χιλιόμετρα σύνορα με τη Συρία, σχεδόν 3 εκατομμύρια πρόσφυγες. Δεν μπορούμε λοιπόν να προβλέψουμε το γεγονός ότι έχουν ισχυρά συμφέροντα ε, και του ενδιαφέρει ιδιαίτερα ε, η κατάσταση της Συρίας. Προτεραιότητα είναι αυτή τη στιγμή το ζήτημα των Κούρδων και η μη ομοιομορφία των τριών περιοχών που βρίσκονται ε, των παραμεθόρων περιοχών. Αλλά για να είμαι ειλικρινή, πιστεύω ότι χωρίς την Τουρκία και τη συμμετοχή της και πολιτικά ακόμη θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια σταθερή λύση για τη Συρία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και τη δική του συμμετοχή, την ενεργό του συμμετοχή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τους 250.000 ανθρώπους στο Χαλέπι, 275.000 ανθρώπους που απειλούνται να γίνουν μετανάστες αυτή τη στιγμή πρόσφυγες, πού θα πάνε. Δεν θα πάνε νότια, θα πάνε βόρεια, στα τουρκικά σύνορα και η Τουρκία, την Τουρκία τη συμφέρει να μην συμβεί αυτό. Αυτό πρέπει να το λάβουμε λοιπόν υπόψη. Έχουμε ήδη επιπτώσεις ε, από την εκλογή του Πρόεδρου Τραμπ. Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, όπου φεύγουν ο Πρόεδρος Ομπάμα και ο Τζον Κέρι. Ε, μέχρι τότε αυτοί θα ασκούν την πολιτική τον ΗΠΑ και βλέπω ότι ο Τζον Κέρι είναι ιδιαίτερα δραστήριο και πιστεύω θα παραμείνει δραστήριο μέχρι την τελευταία ημέρα ε, για να κάνει προσπάθειε να μειωθεί η βία και να γίνουν προσπάθειε υποστήριξη τη ανθρωπιστική βοήθεια. Μετά από αυτά θα χρειαστεί να ξανασυζητήσουμε μεταξύ μα αφού θα γνωρίζουμε ποια θα είναι η ομάδα του Τραμπ και ποια θα είναι η στρατηγική του Τραμπ ε, σε σχέση με τη Ρωσία. Αν θα ακολουθήσει αυτά που ισχυρίζεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του, του Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εστιάστηκα λίγο στα Ηνωμένα Έθνη. Εγώ, ξέρετε, είμαι Ιταλοσουηδός, Ευρωπαίος, ε, έχω Βελγίδα ε, σύζυγο και θέλω η Ευρώπη να υποστηρίξει τα Ηνωμένα Έθνη. Και τα έχετε υποστηρίξει. Φυσικά, εγώ προτεραιότητα θα έδινα στην ανθρωπιστική βοήθεια, διότι εκεί μπορούμε να κάνουμε διαφορά αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, σε επαφή με τις ε, περιφέρειες οι οποίε ακούν τις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά προσπαθεί να κάνει η Φρεντερίκα Μογκερίνη για να διευκολύνει τις επαφές ώστε να κατανοήσει καλύτερα ποια είναι η ατζέντα του για το μέλλον της Συρίας. Υποστηρίζοντα τα όσα κάνουμε εμεί, όχι αντικαθιστώντας τα, γιατί την εντολή την έχουμε εμείς, αλλά υπάρχει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο στα χέρια της Ευρώπης και ονομαστεί ανοικοδόμηση. Γιατί, διότι όλοι, μόλι ανέφερα τη Ρωσία, όλοι στη Συρία και αλλού περιμένουν τη στιγμή όπου ουσιαστικά θα τελειώσει ο πόλεμο για να δουν ποιο και πώ θα ανοικοδομήσει τη Συρία. Αν η Ευρώπη λοιπόν χρησιμοποιήσει τη δική της δύναμη που είναι υπαρκτή ε, και τα συμφέροντά της. Γιατί είναι φθηνότερο να νοικοδομήσει κανείς τη Συρία παρά να απορροφήσει 10 εκατομμύρια ε, πρόσφυγες. Ε, το όφελος θα είναι τεράστιο, αλλά υπό έναν όρο, ότι θα αξιοποιηθεί. Δηλαδή να πει η Ευρώπη να είμαστε έτοιμοι να νοικοδομήσουμε τη Συρία, αλλά μόνο εάν και όταν υπάρξει οικονομική, χωρί αποκλεισμού αξιόπιστη νέα μορφή διακυβέρνηση στη Συρία και όχι απλά μια στρατιωτική νίκη. Αλλιώ χτίστε την μόνη τη Συρία. Α δούμε αν μπορείτε να το κάνετε. και μετά χρωστάω και κάτι στα Ηνωμένα Έθνη, όπου εργαζόμαι εδώ και 46 χρόνια. Έχω χάσει πολλούς συναδέλφους και φίλους στη διάρκεια των διαφόρων 82 φίλους ε, στη διάρκεια της αντιμετώπισης των διαφόρων ε, καταστάσεων, εμπόλεμων καταστάσεων. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας διακόψα, αλλά από ό,τι ξέρετε, οι δερμηνείς μας άντεσαν 18 λεπτά επιπλέον από το χρόνο τους. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα συνεχίσει στις 2.30 τη συνεδρίαση. Ξεκινάμε πιο νωρίς λοιπόν και η Επιτροπή Ανάπτυξη στι 3 εκεί που ήμασταν και κλεισμένο το θηρόν. Σα ευχαριστώ πολύ και καλό διάλειμμα.